Allora, buongiorno a tutti, bentornati. Iniziamo subito come anticipato ieri. Καλημέρα σας. Ας ε, ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας ώστε να προχωρήσουμε στα σημεία που μας μείναν από χθες, το 11 και το 12, συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα. Ε, πακέτο ποιότητα, έτσι το έχουμε αποκαλέσει αυτό εδώ. Η Ράση Γαρσία Πέρες θα μας θυμίσει ε, περί τίνο πρόκειται και πού βρίσκεται η κατάσταση. Θα μπορούσαν να υπάρχουν καινούργιε πράγματα, ε, καινοτομίε. Να μας πει λοιπόν η Ράτζη τι πρόοδος έχει σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες και έπειτα θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όλοι μαζί παρέα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, όντω θα μπορούσα πολλά να σας ε, πω για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Πάντως, η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής. Είναι μια κατάσταση όπου ως Επιτροπή και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρουμε μια θέση. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ, το πακέτο αυτό ποιότητας, έτσι το ονομάζουμε ποιότητας, έχει το σύστημα ποιότητας που από την αρχή των τριμερών διαλόγων το Συμβούλιο επέμεινε για εντολή προς διαπραγμάτευση. Δεν φτάσαμε να το έχουμε συζητήσει στον τριμερή διάλογο, οπότε η πρόταση που κάνουμε εμείς είναι αυτή που κάναμε και σε συμφωνία με τους κοιόδες εισηγητές και είναι όλο το περιεχόμενο της απόφασης που παίρνουμε στην Επιτροπή Γεωργίας για το μάρκετινγκ και τις προδιαγραφές μάρκετινγκ να το προωθήσει και ο εισηγητής, ο κύριος Βαντάν, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης για την κοινή γεωργική πολιτική και στα πλαίσια αυτά να γίνει η συζήτηση επί του περιεχομένου αλλά να ακολουθήσει τη θέση που έχουμε πάρει εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Όσον αφορά τώρα τα συστήματα ποιότητας, οι διαπραγματεύσεις έγιναν και κράτησαν ε, πολλούς μήνες, ένα χρόνο σχεδόν από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα από τα βασικά θέματα για την Επιτροπή μας ήταν αυτό που έχει να κάνει με τον έλεγχο των ε, ποσοτήτων, των όγκων από πλευράς των οργανώσεων των παραγωγών. Ήταν ένα θέμα που μέχρι την τελευταία στιγμή ε, για μας παρέμεινε σημαντικό και επιμείναμε γιατί θέλαμε να υπάρξει συμφωνία. Όμως δυστυχώς έχουμε πάρει αρνητική απάντηση από το Συμβούλιο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Αρνητική στάση βάσει μιας πολιτικής δήλωσης από το Συμβούλιο έχουμε πάρει επίσης προκειμένου το θέμα αυτό να συζητηθεί στα πλαίσια της ε, συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Άρα, Για τα άλλα ζητήματα, εκτός από κανένα δύο θέματα, το πράγμα έχει κλείσει, η συμφωνία έχει κλείσει. Πετύχαμε ως βασικό ζήτημα για την Επιτροπή μας το θέμα που έχει να κάνει με τα προϊόντα από ορεινές περιοχές. Αυτό έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία. Και κάποια άλλα θεματάκια που είναι βέβαια πιο τεχνικά και τα οποία βελτιώνουν το παρόν σύστημα και μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά υπάρχουν δύο τρία ε, πράγματα που ακόμα μας απασχολούν. Φαντάζομαι στις 6 Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το θέμα όταν θα έχουμε τη συνεδρίαση με τους σκιώδες εισηγητές. Ελπίζω τότε να κλείσουν και αυτά τα θεματάκια που παραμένουν. Οπότε τότε στις 20 Ιουνίου θα υπάρξει τριμερής διάλογος και η ιδέα θα είναι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία με την ε, Προεδρία της Δανίας στις 25 Ιουνίου. Πάντως, η θέση που υποστηρίζουμε δεν είναι μόνο δικιά μου, της εισηγήτριας, είναι μια συμφωνία την οποία στηρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες, πρέπει να ξέρετε. Και όταν έπρεπε να επιλέξουμε είτε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και άρα να πάμε σε δεύτερη ανάγνωση ή να πετύχουμε συμφωνία βάσει πολιτικής συμφωνίας, όπως σας είπα πριν, κατά πλειοψηφία αποφασίσαμε να διαπραγματευτούμε και να πετύχουμε συμφωνία, παρόλο που όλες οι πολιτικές ομάδες δεν είχαν την ίδια άποψη. Κατά πλειοψηφία αποφασίσαμε. Όπως είπα, πρόκειται για μια προσπάθεια που κάνουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να κλείσουν ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν και στις 25 Ιουνίου η Ποδανέζικη Προεδρία να υπάρξει πολιτική συμφωνία για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, καλώς. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, μας δείξατε το δρόμο. Αυτό το δρόμο λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί όσον αφορά τις ποσότητες. Κύριε Ντόρφμαν, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ιράτσε για την εργασία της. Το είπε και εκείνη ότι ενημερωνόμαστε τώρα για αυτό το θέμα και μάλιστα έχουμε επιτύχει ένα σωρό θετικά πράγματα. Ωστόσο, Ορισμένοι όμιλοι όπου η κύκλη εργασιών είναι πολύ ψηλή και όμιλοι που ασχολούνται με προϊόντα όπου η ορίμαση παίρνει χρόνο, δηλαδή η περίοδος από τότε που αποφασίζει κανείς να παράγει μέχρι να πωλήσει είναι πολύ μακρά, Εκεί ο καθορισμός των όγκων θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι κάπως παράξενο. Και στο γάλα φτάσαμε σε συμβαστική λύση ε, με το Συμβούλιο αλλά και για το τυρί ε, που με μακράς ε, ορίμανση το ίδιο αλλά για τα υπόλοιπα δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. και εμείς στο εσωτερικό της πολιτικής μου ομάδας έχουμε συζητήσει επί μακρόν πώς θα προχωρήσουμε και τη γνώμη μου αν θέλουμε να τελειώνουμε τώρα στην πρώτη ανάγνωση με το αποτέλεσμα που έχουμε φτάσει δηλαδή χωρίς προγραμματισμό δύο πράγματα πρέπει να τα πούμε. Καταρχήν χρειάζεται αυτή η πολιτική δήλωση από το Συμβούλιο, που το Συμβούλιο σημειώνει και διαπιστώνει ότι αυτό το, σύστημα, αυτό το επιχείρημα είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Και έπειτα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αμέσως πώς θα εξετάσουμε αυτό το επιχείρημα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Διότι είμαι πεπισμένος ότι είναι χρήσιμο να ενταχθεί αυτό το επιχείρημα εκ νέου στον κανονισμό της ενιαίας ΚΟΑ και να ξαναρχίσουμε αυτού και από την αρχή ελπίζοντας ότι το Συμβούλιο αργά ή γρήγορα θα το δεχτεί και θα βρούμε μια λύση. Καλύτερα είναι λοιπόν να κλείσουμε τώρα στην πρώτη ανάγνωση για να σιγουρέψουμε τα όσα έχουμε πετύχει που σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Χέρμπερτ. Πολύ σαφή η θέση σου. Και τώρα δίνω το λόγο στο Σμιτ και μετά στο Ρέιμερς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρέπει να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε συγχαρητήρια στην Αράντσα. Ήταν πραγματικά περίπλοκες οι διαπραγματεύσεις και πολύ σύνθετες και σίγουρα δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα. του λεχθέντος έχουμε και τα στοιχεία όσον αφορά και το Συμβούλιο και την Πολιτική όσον αφορά την Επιτροπή μας. Κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Αλλά πρέπει η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή να γνωρίζει ότι ακόμα και αν ε, δίνουμε πράγματι μια προοπτική για αυτό τον γενναίο νέο κόσμο και για την αξιοπρέπεια όσον αφορά το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο, σε σχέση με όλες τις διαπραγματεύσεις κάναμε ό,τι μπορούσαμε αλλά δεν ήθελε, δεν κατάφερε το Συμβούλιο να πιστεί και δεν κατάφερε, δεν ήθελε καν να κινηθεί. Και έτσι μας έδωσε ψίχουλα, στο το πω έτσι. Το γεγονός ότι πολιτικές δηλώσεις από κάποιους πολιτικούς δεν αξίζει και πολλά πράγματα όσο ακριβώς και η αρχική θέση για τη διαπραγμάτευση είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικός ο τρόπος αυτός λειτουργίας σε σχέση και με τα αποτελέσματα. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να εργάζεται και να πετυχαίνει το Κοινοβούλιο τόσο ισχνά αποτελέσματα. Πρέπει να καταφέρουμε να είμαστε πιο επιτυχείς. Υπάρχει πλειοψηφία σε σχέση με τις ομάδες για αυτά τα θέματα. Επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να καταθέσουμε τροπολογίε στην Ολομέλεια. Ήταν αξιοθρύνητη η τοποθέτηση, η θέση του ε, θεσμικού μας οργάνου. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Είναι πραγματικά απογοητευτική θετική αυτή η κατάσταση για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ. Δεν έφτασε ακόμα ο Μισελ Ντεντάν, αλλά Όπω ξέρει καλά ο εισηγητή και οι σκιάδες εισηγητέ, έχει ήδη φροντίσει να συμπεριλάβει αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας, δηλαδή τη ρύθμιση των όγκων στην ενιαία ΚΟΑ. Μπρίτα Ρέμερς. Ε, ουσιαστικά δεν μένουν πολλά να πω, έχουν αναφερθεί τα περισσότερα. Καταδεικνύεται για άλλη μια φορά όμως ότι η κατηγορία ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο είναι λέει το φρένο που έχει τραβήξει, τροχοπεδί τα πράγματα για τις διαπραγματεύσεις δεν αληθεύει. Επανειλημμένα το Συμβούλιο τροχοπεδεί τα πράγματα. Δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε αποτελέσματα από τι διαπραγματεύσει. Δεν υπάρχει αρκετή εντολή, α το πω έτσι, εύρο εντολή για να προχωρήσει και καταδεικνύεται ότι όλα σε πρώτη ανάγνωση είμαστε υποχρεωμένοι να τα επιλύσουμε, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν μπορούμε διαρκώς να υπαναχωρούμε επειδή μπορεί πιο εύκολα έτσι να συμφωνεί, λέει το Συμβούλιο. Πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε εσωτερικά, για να υπάρχει μια εσωτερική συμφωνία, αλλά δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό το Συμβούλιο. Εξού και νομίζω τώρα ήρθε η χρονική στιγμή να βρούμε μια άλλη πορεία, να μην είμαστε κατακαιρματισμένοι. Αναμένω να δω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.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 nel proseguire questo lavoro. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται διαγράφεται μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της συνέχισης της εργασίας της συζητήτης. Φυσικά θα συνεχίσουμε την μάχη, όπως δεν υποχωρήσαμε στο πακέτο για το γάλα, δεν θα υποχωρήσουμε ούτε και για το πακέτο για την ποιότητα. Θέλουμε όμως να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα και εγώ θέλω μόνο ένα από αυτά να θυμίσω σε αυτόν τον κανονισμό για την ποιότητα των κανόνα εξοφίτσο που είναι πολύ μεγάλη ε, πολύ μεγάλη σημασία για το Κοινοβούλιο, όχι μόνο γιατί συμφωνούμε, αλλά γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ε, ισχυρό όπλο στην προστασία της ποιότητας, των προϊόντων ποιότητας τα προϊόντα των ορνών περιοχών. Είχαμε κάνει έναν αγώνα γι' αυτό. Η Κομισιόν δεν το είχε εισάγει. Τώρα το δέχτηκε. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια σαφή πολιτική δήλωση που θα λέει, θα διευκρινίζει μάλλον ότι ο ρόλος μας ως Επιτροπή Γεωργίας είναι να προχωρήσει η καταγραφή των προϊόντων αυτών. Θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι το Συμβούλιο δεν έχει πετύχει ε, πλειοψηφία όσον αφορά τον έλεγχο των όγκων. Εάν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, η Ράτζη προχώρη και πες μας για το τι έγινε με τη συνεδρίαση της 20ης και της 25ης ε, και να δούμε αν θα μπορέσουμε ε, να κλείσουμε τη συμφωνία και να περάσουμε γρήγορα και στο σημείο 12, γιατί υπάρχει ακόμα μια σημαντική, ε, ένα σημαντικό νέο. Διακόπτει Πρόεδρος. Eh, modifica Τροποποίηση του κανονισμού 73 ε, ε, του 2009 ε, άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς. Εδώ το συζητήσαμε στο Στρασβούργο. Να ρωτήσω λοιπόν τον Λουίση να με ενημερώσει την Επιτροπή μας για τα νέα μετά από τον τριμερή διάλογο. Λουίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρόκειται για μια έκθεση εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά τη σταθερότητα που είναι απαραίτητο να δοθεί στους ε, γεωργούς για το 2013 από τη στιγμή δηλαδή που η σημερινή προγραμματική περίοδος από την άποψη την δημοσιονομική κλείνει το 2012 άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να αγγιηθούμε τη μετάβαση για το 2013 που δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην ε, ομαλή εξέλιξη των γεωργικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πρόταση με την οποία, τη βάση της οποίας δουλεύουμε αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορούσα παρά να αναφέρω την ξέρετε συνεργασία που είχα με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Θέλω να, τους χαιρετήσω, να χαιρετήσω όλους την κυρία Κριστίνα Μπόρσμαν και την ομάδα της, το επιτελείο της που μας έδωσε από την τεχνική άποψη πολύτιμη βοήθεια, καθώς ακόμα και ολόκληρη την, την Επιτροπή, συγγνώμη, την Γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας. Ε, κάναμε μια άτυπη τριμερή επαφή στο Στρασβούργο. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί η Κομισιόν δέχτηκε όλες μας τις προτάσεις ε, που συνήθως αντιστέκεται σε αυτές. Πιστεύω πως αυτό είναι ένα καλό σημάδι ε, για τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για τις υπόλοιπες εκθέσεις, αλλά όλα αυτά σημαίνουν και ότι θα μπορέσουμε σύντομα να λύσουμε το πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, τέθη ένα νέο θέμα, χρειάστηκε να αλλάξει η νομική βάση για να καλύψουμε συγκεκριμένα προβλήματα κάποιων κρατών μελών. Και τι, τι σημαίνει, σημαίνει η αλλαγή μας ότι πρέπει να πάρουμε τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα, αυτό μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία και με όλη αυτή την καθυστέρηση μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό που όλοι επιθυμούμε, δηλαδή την ταχεία έγκριση αυτού, αυτής της έκθεσης, έτσι ώστε το δημοσιονομικό έτος χρήση 2013 να μην έχει προβλήματα. Η Γερμανία ε, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και κράτη, νέα κράτη-μέλη ένα σύνολο συγκεκριμένων προβλημάτων με πολύ περίπλοκες επιπτώσει, που με αυτή τη μορφή είναι εύκολο είναι δυνατόν να λυθούν και ελπίζω πως τώρα εντό του Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να συντομεύσουμε όσο γίνεται τις προθεσμίες και ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο αν είναι δυνατόν να έχουμε μια άμεση και προσωπική επαφή με τον συνάδελφό σας, ε, τον ομόλογό σας της Επιτροπής ε, της Νομικής, ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, να περάσει ήδη από την Ολομέλεια, αν γίνεται και τον Ιούλιο. Ο Σεπτέμβριος είναι ένα όριο και ήδη μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα, αλλά πάντως ε, βασικά αυτά είναι τα θέματα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που επέβαλαν τροπολογίες και να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά την Κομισιόν και την Γραμματεία για τη βοήθεια που προσέφεραν ώστε να ολοκληρωθεί αισίως η εξέταση αυτού της έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα ένα σημαντικό σημείο. Παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι έχουμε τουλάχιστον τρεις θέσεις στις οποίες θα πρέπει να είμαστε σήμερα το πρωί. Όταν λέμε ψηφίζουμε σε νέα, πρέπει να ψηφίζουμε σε νέα. Και επειδή για τους σοσιαλιστές ε, ε, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιοι καθυστέρησαν και δεν ήρθαν, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλους τους σοσιαλιστές ε, εισηγητές για να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο. Ας ξεκινήσουμε και με τις ψηφοφορίες. Όταν λέμε νέα όπως είχε προαναγγεθεί έτσι πρέπει να γίνεται. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω ότι χτες ε, αλλάξαμε την ε, σημερινή μερίσια διάταξη και ακολουθούμε αυτά που αποφασίστηκαν. Ε, τότε πρέπει να ενημερώνετε όμως τους ε, βουλευτές, παρακαλώ. Ναι, ναι. Πρέπει να το ενημερωθήκατε από χτες το μεσημέρι που ψηφίσαμε την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. allora col 7 σημείο 7 τη της διάταξη. Παρακαλώ όλοι να πάρετε τι κάρτε σα ψηφοφορία. Έκθεση λοιπόν για το εντολή για τον τριμερή διάλογο. Έστε τελάν και 14 τροπολογίε έχουν υποβληθεί. Θα ήθελα να θυμίσω στα μέλη τη Επιτροπή ότι έχουμε προθεσμία για τα αιτήματα για τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσει τη 4η Ιουνίου. Το αργότερο. Allora, possiamo iniziare la votazione. Budget, yeah. Ok. Aperta la votazione sul punto 1. Άρχεται η ψηφοφορία για το σημείο 1. Τροπολογία 1. Ρόντουστ. Απέρτα la votazione. No, it doesn't work. It doesn't work. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, δεν δουλεύει. Α, τώρα δουλεύει. Τώρα λειτουργεί. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Τροπολογία 1. Ε, απορρίπτεται. 2. Ψηφίζουμε για τη 2. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για τη συμβιβαστική 1. Συμβιβαστική 1. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας για τη συμβιβαστική 1. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6. Λάιον και λυπή. Τέλος της ψηφοφορίας. Τροπολογία 6. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 7. 7. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 9. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Adesso apro la votazione sul numero 8. Votiamo. Τώρα ψηφίζουμε για την 8 Νικουλέσκου. Ε, ψηφίζουμε τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 10 Ashworth. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 12, Λάιον και άλλοι. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 11. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τέλος 14. Ψηφίζουμε για τη 14. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα έχουμε στο σημείο 6 ακόμα μια ψηφοφορία. Συνάδελφοι. Πρόεδρε, μια παράκληση έχω. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη βέβαια στην δική σας αξιολόγηση για την ψηφοφορία. Δεν μπορούμε όμως να δούμε πώς συγκεκριμένα ψηφίστηκε. Και τουλάχιστον να γνωστοποιείτε παρακαλώ ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας. Όχι ότι αμφιβάλλω γι' αυτό, αλλά αν είναι 18-7 δεν το ξέρουμε ή 18-13 δεν το βλέπει κανείς από την οθόνη. Ίσως θα μπορούσατε να το βάλετε ή να το πείτε. Ευχαριστώ. Αν νόμιζα πως ε, άναβε στον πίνακα. Εντάξει, θα το, φροντίσω. Άγνιου. Ζητώ συγγνώμη σας καθυστερώ. Εγώ ψήφισα λάθος την πρώτη ψηφοφορία. Δεν θα είχε κάνει διαφορά. Έπρεπε να είχα ψηφίσει όχι και ψήφισα ναι. Mm, ε, εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα, αλλά θα καταγράψουμε την αρνητική σας ψήφο. Ωραία. Ξεκινάμε με το σημείο 6, την δημιουργία ενός δικτύου λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο εισηγητής ο Τζαν Κάρλο Σκοτά. Και εδώ λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ο Σκοτά λείπει. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο, πάντως θα κάνουμε την ψηφοφορία. Μάλιστα. Ψηφίζουμε. Λοιπόν, τροπολογία 1. Τέλος της πληροφορίας. Εντάξει, Πέτερ, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα. Τέλεια. Ωραία. Όλοι είναι ευχαριστημένοι, αλλά και ανήσυχοι. <laughs> Γέρεμιστε λίγο. Λοιπόν, σημείο 3. Νατελτσέβα. Ψηφίζουμε τέλος ψηφοφορίας. Έγκρινατε. Τροπολογία 4 που λέει να ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες 6 μέχρι και 10. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Οι 4, οι 6 και οι 10 λοιπόν εγκρίθηκαν. Πάμε στην 5 λοιπόν. 5. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 5. Μπρίτα όμως θέλει λίγο το λόγο. Ε, Δεν θέλω να μακρηγορήσω για την δική μου τροπολογία από την νομική υπηρεσία υπήρξαν κάποιες τροποποίησεις. Ε, η πρόταση κάπως αναδιατυπώθηκε, ας το πω έτσι, ώστε να ταιριάζει με το άρθρο 290. Και γι' αυτό θα λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εξουσία να δώσει εντολή για κατεντολήν, κατεξουσίαν πράξη σύμφωνα με το άρθρο αυτό για τον σκοπό τροποποίησης μετά από έτοιμα κράτου μέλους του καταλόγου που θα ε, αναφέρεται στις επιδοτήσεις ενισχύσει κρατικές. Είναι μια αναδιατύπωση αυτή, είναι σαφές. Va bene. Grazie Britta. Apriamo Μάλιστα, ευχαριστώ Μπρίτα. Ψηφίζουμε για τροπολογία 5. Τέλος της ψηφοφορίας. Γκρινεται. Τροπολογία 8. Ashford. Άρχεται η ψηφοφορία. 8. 8. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Adesso apriamo la votazione sull'emendamento. Και τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 9. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίφθηκε και η 9. Πάμε τώρα για την 2. Ψηφίζουμε την 2. Τροπολογία 2 του εισηγητή. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση έτσι όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε για την νομοθετική πρόταση. Εγκρίνεται λοιπόν. Και τώρα για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητηρία στον εισηγητή Τζαν Κάρλο Σκοτά και μπορούμε να προχωρήσουμε. Τελειώσαμε με το 6 και με το 7 και μπορούμε να πάμε στο 8. Ποιος πήρε το λόγο? Ο Μάγερ, παρακαλώ. Bravo. Για αυτό το τελευταίο σημείο μία παρατήρηση ακόμα για την τελευταία ψηφοφορία. Οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο δεν θα είναι απλέ ω εγχείρημα, γιατί έχουμε το παλαιό πρόβλημα εδώ μπροστά μα. Θέλει να έχει κατεντολήν εξουσιοδότηση για πράξει ε, το Συμβούλιο, ενώ θέλει εκπροσωπ... εκπροσωπούμενε πράξει στο Κοινοβούλιο και έχουμε, βλέπετε το θέμα αυτό λόγω του κανονισμού των ρυθμίσεων. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν σε αυτές, σε αυτές τις Ευρωκοινοβούλιο. Δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε. Οι κανονισμοί είναι ε, εκπροσωπούμενες πράξεις και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Μάγερ, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και λεπτό. Να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι για αυτό το σημείο λάβαμε μια επιστολή πολύ συγκεκριμένη ως πρόεδρο της Επιτροπής, ως πρόεδρος της Επιτροπής από τον πρόεδρο Λένε που είναι ο πρόεδρος του Συνόλου των Προέδρων των Επιτροπών και για να μην διατρέξουμε το κίνδυνο να μην φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία για τα σημαντικά θέματα, να υποβαθμίσουμε τα σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την εφαρμογή, δηλαδή της κατεξιοδότηση πράξης ή τις εφαρμοστικές ε, διατάξεις. Τον Ιούλιο λοιπόν στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τις πράξεις τις οποίες θα έχουμε συζητήσει με το Συμβούλιο Επιμακρών όσον αφορά την ευθυγράμμιση με τη Λισαβόνα για τις άμεσες πληρωμές, την, ε, ανάπτυξη, την ε, ανάπτυξη της υπέδρου και την ενιαία ΑΚΟΑ και Εκεί όπου δεν έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο θα σημειώσουμε την δική μας αντίθεση με αυτή την ψηφοφορία στην Ολομέλεια που ελπίζω θα είναι πολύ σημαντική ε, και από εκεί θα ξεκινήσουμε κύριε Μάγερ όπως μας καλεί να το κάνουμε η Επιτροπή. Δεν κάνουμε καθόλου πίσω. Σας ευχαριστώ και περνάμε στο σημείο 8. Τώρα, colleghi, un minuto solo di interruzione, sta arrivando... Ένα λεπτό διακοπή θα κάνουμε. Φτάνει ο εισηγητής Ρενέ Σουσόν από την Επιτροπή Περιφερειών. Μόλις μπει θα ξεκινήσουμε. Mm. So, so, so,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 che ci ha raggiunto. Ξαναξεκινάμε με την παρουσία του κυρίου Ρενέ Σουσό και να του δώσουμε το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεση και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Merci, euh, Monsieur le Président. Bonjour à toutes Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ. Η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθέτησε την γνωμοδότηση που σας υπέβαλα στις 4 Μαΐου με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Μόνο τρεις ψήφοι κατά υπήρξαν. Συνεπώς θα σας μιλήσω για τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο πυλώνα και πιο συγκεκριμένα για την αγροτική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση. Ποιοι είναι οι άξονες της δικής μας πρότασης. Σίγουρα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν ε, καλοί προσανατολισμοί. Όμως, όμως βρισκόμαστε πολύ μακριά από μια σε βάθο μεταρρύθμιση η οποία θα μας επέτρεπε να φτάσουμε και να πετύχουμε τους στόχους που καθορίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων σημαντικών στόχων είναι μια γεωργία σε ολόκληρη την επικράτεια. Όμως οι προτάσεις δεν μας επιτρέπουν να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ένας άλλος ε, στόχος ήταν η συμμεταχείριση όλων των γεωργών. Ένα επίπεδο ζωής συγκρίσιμο με το σύνολο της κοινωνίας. Κάθε φορά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι προσανατολισμοί είναι μεν καλοί και σωστοί, τα μέσα όμως που διατίθεται για την επίτευξή τους δεν επαρκούν. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Ποιες είναι οι κυριότερες αδυναμίες. Πρώτα απ' όλα η ρύθμιση ή μάλλον η έλλειψη ρύθμισης των αγορών. Οι μηχανισμοί που προτείνονται είναι μηχανισμοί για θεραπεία όταν υπάρχει κρίση. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόληψη. Αντίθετα, υπάρχει η κατάργηση όλων των ρυθμιστικών διατάξεων που έδειξαν ότι αξίζουν. Είτε είναι οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, είτε τη ζάχαρης, είτε της αμπέλου κτλ. Γι' αυτό και η Επιτροπή των Περιφερειών θα ήθελε ακριβέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάργησης αυτής. Κυρίως των μηχανισμών για την διαχείριση της κρίσης που δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση των εισόδων των γεωργών. Αν δεν υπάρχει ρύθμιση τότε κάθε γεωργός σε όσο πιο δύναμη θέση βρίσκεται τόσο μεγαλύτερα προβλήματα θα έχει. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο τροφοδοτεί τη συζήτηση στον τύπο για παράδειγμα είναι η οροφή και η φθήνουσα κατάσταση, η μείωση δηλαδή σταδιακή. Όσον αφορά την οροφή, πάει πιο μακριά από αυτό που θέλει η Επιτροπή. 200.000 αντί για 300.000 που προτείνει η Επίτροπη και μια φθήνουσα κατάσταση πιο σταδιακή. Κατά τη γνώμη μου, και εξάλλου είναι πολύ ευαίσθητα σε αυτό τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, είμαστε πολύ επικριτικοί όταν βλέπουμε ποιος παίρνει τελικά την βοήθεια. Ο μέσος όρος της βοήθειας το 2000... 2011 ήταν 5.093 ανά εκμετάλλευση. Και τι λέμε, δεν πρέπει να υπάρχει όριο. Έχετε 3.970 εκμεταλλεύσεις. Το 2010, που πήραν δηλαδή το 2010, πάνω από 300.000 ευρώ. Η διαφορά είναι μεγάλη. Και πίσω από όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι κοινωνικά οι ενισχύσεις αυτές ε, δύσκολα γίνονται αποδεκτές, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα οικονομικά προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε ορισμένες χώρες πάρα πολύ μεγάλα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε από δημόσιο χρήμα ποσά τόσο υψηλά Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή των Περιφερειών είναι, κατάλαβε πάρα πολύ καλά τη δικιά μου την πρόταση και θέλει την οροφή που στα 200.000 ευρώ βάζει μέσα το μέτρο του 30% ε, για το πρασίνισμα της Γεωργίας. Κάτι άλλο τώρα. Η σύγκληση. Η σύγκληση των ενισχύσεων, όχι μεταξύ των μέσα στις χώρες μάλλον, γιατί οι χώρες το καθορίζουν αυτό, αλλά διακρατικά. Βλέπετε πολλές χώρες ότι έχουν επίπεδα τα οποία δεν είναι καθόλου στο ύψος των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Οι βαλτικές χώρες, για παράδειγμα. Και γενικά οι νέες χώρες. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια πολύ γρήγορη σύγκληση, να προβλέψει παρόλα αυτά ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, διακρατική σύγκλησης με συγκεκριμένα κριτήρια. Γιατί αν βασιζόμαστε σε μία ενίσχυση ανεκτάριο που είναι η ίδια παντού, ε, δεν στέκει οικονομικά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος της παραγωγής και άλλες παραμέτρους. Πάντως το θέμα αυτό πρέπει να το δουλέψουμε. Γιατί η σύγκληση είναι αναγκαία τελικά. Άρα η θέση μας είναι ισορροπημένη γιατί ζητάμε χρονοδιάγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα εφαρμοστεί. Τώρα όσον αφορά τη σύνδεση των ενισχύσεων. Η Επιτροπή των Περιφερειών πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή η σύνδεση, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν δυσκολίες λόγω της φυσικής τους κατάστασης, δηλαδή νορινές, απομακρυνμένες κτλ. Η γεωργία ιδεολογική επίσης πρέπει να προωθηθεί και η γεωργία ποιότητας, η οποία πρέπει να υποφεληθεί από τα μέτρα αυτά. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο πολύ επίμαχο σημείο. Και αυτό είναι το πρασίνισμα της Γεωργίας. Υπάρχει μια πρωτότυπη πρόταση από την Επιτροπή των Περιφερειών. Όλοι συμφωνούν για το ότι τα μέτρα αυτά πρασινίσματος, το 30% δηλαδή, δεν μπορεί ομοιόμορφα να εφαρμοστούν παντού. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη διαφοροποίηση της καλλιέργειας, τα αγρονομικά χαρακτηριστικά, το μέγεθος κλπ. Χρειάζεται δηλαδή κάποια ευελιξία ε, στα μέτρα αυτά. Παρόλο που ο στόχος παραμένει να προχωρήσουμε προς την αηφόρα ανάπτυξη, προς την βιώσιμη γεωργία. Το 30% δεν είναι πρόβλημα για μας. Αυτό που είναι πρόβλημα για μας είναι η εφαρμογή που κινδυνεύει να γίνει υπερβολικά ομοιόμορφα και άρα με άκαμπτο τρόπο. Τα μέτρα λοιπόν που προτείνουμε και που έχουν να κάνουν και με το 30% και με το 7% της οικολογικής επιφάνειας είναι το λάβουμε υπόψη μας πώς διάφορες μικρές ε, επιφάνειες θα μπορούσαν να μπουν μαζί. Να υπάρξουν δηλαδή κάποιες, κάποιοι εταιρικέ σχέσεις, συνεταιρισμοί μεταξύ γεωργών και ε, περιφερειών ή τοπικών αρχών. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γίνει αυτό και έτσι έχουν μπει οι επιφάνειες αυτές οι βιολογικές όλες μαζί για να καλύπτεται αυτό το 30% που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε δηλαδή σε μια συγκεκριμένη περιοχή να το πετύχουμε αυτό και να δεχτούμε ότι για μια εκμετάλλευση να είναι 3% αλλά σε μία άλλη να έχουμε 12-13%. Καταλάβατε, να τα βάλουμε αυτά μαζί και να έχουμε ένα μέσο όρο που να αντιστοιχεί στο 7%. Να μην δυσκολέψουμε δηλαδή υπερβολικά τους γεωργούς. Για τις ε, περιφέρειες λοιπόν που λόγω της φυσικής τους κατάστασης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα ορεινές κλπ. Εδώ τα μέτρα πρέπει να είναι υποχρεωτικά κατά τη γνώμη μας για τις διάφορες χώρες και όχι σε θελοντική βάση. και να μπορούν να πάνε μέχρι και 10% από τον πρώτο πυλώνα στις ε, περιοχές αυτές εφόσον θέλουμε να διατηρηθεί εκεί η γεωργική δραστηριότητα. Για τις εγκαταστάσεις τώρα. Ε, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση για να ευνοηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις και θέλουμε να υπάρξει και η έννοια της νέας εγκατάστασης. Δηλαδή όχι μόνο η έννοια του νέου γεωργού, αυτό το έχουμε από παλιά με όριο τα 40 χρόνια. Κάτι το οποίο όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά που δεν είναι κάτω από 40. Αντί για την έννοια λοιπόν του νέου γεωργού να βάλουμε την έννοια του, της νέας δραστηριότητας, του ατόμου που εγκαθίσταται για πρώτη φορά και αναλαμβάνει μια τέτοια δραστηριότητα. Έρχομαι στο δεύτερο πυλώνα τώρα. Ανάπτυξη της υπαίθρου. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι εφόσον δεν υπάρχει ρύθμιση της αγοράς, έχουμε και την μεγαλύτερη απογοήτευση της Επιτροπής των Περιφερειών απέναντι στις προτάσεις της Κομισιόν. Φυσικά και υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, ιδιαίτερα το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τα Διορθωτικά ταμεία και το ΦΕΝΤΕΡ, το Περιφερειακό δηλαδή, Ταμείο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, όπως και η ολοκλήρωση. Δηλαδή το γεγονός ότι εντάσσεται στη στρατηγική 2020 η Γεωργία. Έπειτα ότι το πρόγραμμα Leader μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα ταμεία. Όλα αυτά είναι θετικά. Όμως τα μέσα και πολύ περισσότερο στο δεύτερο πυλώνα από ό,τι στον πρώτο. Τα μέσα, τα κονδύλια δηλαδή, δεν φτάνουν για να έχουμε την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Οι έξι προτεραιότητε τώρα, οι οποίε αναφέρονται στην πρόταση της Κομισιόν, διαρθρώνονται ελάχιστα μεταξύ τους. Στις προτεραιότητες αυτές, οι δυνατότητες αυτές, συμπεριλαμβάνεται μηχανισμός διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με την αγορά είναι κάτι πολύ συμβολικό. Γιατί η διαχείριση του κινδύνου για την γεωργική παραγωγή δεν έχει καμιά δουλειά στο δεύτερο πυλώνα, όπου τελικά βάζουμε λίγο απ' όλα ό,τι θέλουμε να ξεφορτωθούμε από αλλού. Όχι. Η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να είναι αποκλειστικά στον πρώτο πυλώνα. Αποκλειστικά. Για το δεύτερο πυλώνα τώρα πάντα είμαστε ανάμεσα στη γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Η Κομισιόν, τουλάχιστον αυτό συστήνει η Επιτροπή των Περιφερειών, πρέπει να προτείνει μια πραγματική στρατηγική ανάπτυξη τη υπαίθρου. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξη τη υπαίθρου που να προσαρμόζεται σε κάθε χώρα στα πλαίσια των συμβολέων εταιρική σχέση έτσι όπω τα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δικιά μα Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει δύο υποπρογράμματα θεματικά υπέρ της παραγωγής ποιότητας που δεν στηρίζεται αρκετά πρώτον και δεύτερον υπέρ της περιαστικής παραγωγής γύρω από τις πόλεις δηλαδή που υπάρχει σε πολλές ε, περιοχές γιατί μην ξεχνάμε οι πόλεις ζουν, τρέφονται από τις ε, αγροτικές περιοχές από την Ήπεθρο δηλαδή. 10% των κονδυλίων από τον πρώτο πυλώνα λοιπόν θα έπρεπε να μεταφερθεί στο δεύτερο πυλώνα. Βέβαια, οι χώρες μέλη αποφασίζουν. Είναι όμως μια δυνατότητα που είναι ανοιχτή. Θέλουμε να γίνει μια προσπάθεια για την έρευνα και την καινοτομία για την πολιτική της υπαίθρου. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο μου θέμα που είναι η διαχείριση και η εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί, γιατί το πλαίσιο της πολυεπίπεδης διαχείρισης, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δηλαδή, είναι ζωτική σημασία για να διατηρήσουμε την ε, διαφοροποίηση της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου. Η Επιτροπή προτείνει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τη διαχείριση ΦΕΝΤΕΡ, ΦΕΑΜ, ΤΕΦΕΣΕ κτλ. Κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Όμως, για να είμαστε συνεπείς και αποτελεσματικοί, πρέπει τα συμβόλαια εταιρικής σχέσης που γίνονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κάθε χώρα μέλος να ε, έχουν ε, ως στόχο το περιφερειακό επίπεδο. Γιατί έτσι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα μπορούν να χτίζουν την αγροτική και περιφερειακή τους πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βέβαια θα έχουν και τα μέσα στη διάθεσή τους να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους στην πραγματικότητα που ισχύει επιτόπου στη δικιά τους επικράτεια. Στο κείμενο όμως οι τοπικές αρχές αποκλείονται από αυτό το συμβόλαιο κομισιών ε, χωρών μελών. Γι' αυτό και ζητούμε εμείς να συμπεριληφθούν. Ζητάμε επίσης να είναι παρόν και ένας εκπρόσωπος των τοπικών αρχών στην Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Υπέθρου που θα βοηθάει την Κομισιόν στις κατεξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες προβλέπονται όπως γνωρίζετε και πρόκειται να είναι πολυάριθμες. Με δύο λόγια, λοιπόν, αυτό που διακυδεύεται στο νομοθετικό πακέτο που έχουμε είναι η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και η άμεση σχέση των τοπικών αρχών με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειοποίηση της διαχείρισης. Πώς δηλαδή το τοπικό επίπεδο θα συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής. Τέλος, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, όπως προτείνεται, είναι το ελάχιστο και κάτω από αυτό δεν θα έπρεπε με τίποτα να πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, Σουσόν για αυτή την έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών. Τώρα θα έχουμε τη συζήτηση. Ήδη ζήτησε το λόγο ο κύριος Γιάρ και μετά ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πρώτα για τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις και τις συγκεκριμένες επισημάνσεις και προτάσεις. Για μένα η Επιτροπή των Περιφερειών είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή, διότι άμεσα διασφαλίζει την επαφή μεταξύ Ευρωβουλευτών προς την πολλές φορές επενεμένη και σημαντική βάση τι πρέπει να γίνει γεωργικά στην, στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα στις περιφέρειές μας και πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Γι' αυτό οι απόψεις σας και οι γνωμοδοτήσεις σας είναι πολύ σημαντικές για μας. Τρεις-τέσσερις ερωτήσεις θα είχα Πρώτη ερώτηση για τα χρήματα, τα κονδύλια. Στους γεωργούς είναι γνωστό γενικά ότι πρέπει να ταΐσουμε πρώτα την Αγελάδα προτού την αρμέξουμε και εξακολουθούμε να έχουμε έντονες συζητήσεις στα κράτη-μέλη για το ύψος των ε, εισφορών και των συνεισφορών. Είναι ανοιχτή αυτή η συζήτηση. Η Επιτροπή Περιφερειών έχει σημαντική επιρροή στα κράτη-μέλη βέβαια. Ποια είναι η άποψή σα, ποια είναι η άποψή σα συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, ποιο θα έπρεπε να είναι το ποσοστό συμμετοχή, το input, τα κονδύλια από πλευρά εισφορών ε, τη, για την κατανομή αυτών των κονδυλίων πρέπει πιο, πρώτα, πρέπει πιο πριν να τα έχουμε ε, εισπράξει για το πρασίνισμα, greening. Πολλές ιδέες αναπτύξατε που είναι ενδιαφέρουσες. Η ερώτησή μου είναι μια και στην Επιτροπή παρακολουθούμε τις προτάσεις του Επιτρόπου και είπαμε, Επιτρόπου για τη Γεωργία, και είπαμε εντάξει θέλει την Γεωργία για τους πολίτες να την καταστήσει πιο ανοιχτή και πιο φιλοπεριβαλλοντική, πιο πράσινη. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε το θετικό γεγονός ότι σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε πολλά είδη προγράμματα για το περιβάλλον σε θελοντική βάση που υλοποιούνται με τους γεωργούς και δίνουμε αγώνα ώστε αυτές οι εκμεταλλεύσεις, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αυτά τα αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά προγράμματα εφαρμόζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα, αυτές οι εκμεταλλεύσεις να απελευθερώνονται από το πρασίνισμα. Θα ήταν ένα, ε, μια κατάσταση που θα ίσχυε όπως και για τις επιχειρήσεις που είναι οι φιλοοικολογικές. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή την ιδέα. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου, τρίτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι η συγχρηματοδότηση έχει συζητηθεί και έχει οριμάσει αρκετά. Παίρνουμε όλο και περισσότερα μηνύματα από τις περιφέρειες ότι δημιουργούνται όλο και περισσότερα, προβλήματα να συγχρηματοδοτήσουν οι περιφέρειες. Αν αυτό συμβαίνει η ερώτησή μου είναι έχετε κάποιες προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων. Αυτά ήταν οι ερωτήσεις μου. Αυτές ευχαριστώ. Grazie E Dorfman και μετά ο κύριος Ντόρφμαν, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή από την Επιτροπή των Περιφερειών για αυτή τη γνωμοδότηση που πέρσι είχαμε και την ευκαιρία να επισκεφθούμε με την, την περιφέρεια αυτή που είναι μια πραγματικά διαμορφωμένη από τη Γεωργία η περιφέρεια αυτή και διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δύο θέματα θα ήθελα μόνο για άλλη μια φορά να τονίσω, να αναφέρω διότι πρέπει νομίζω στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτά τα θέματα. Το ένα είναι το θέμα της πρόσθετης υποστήριξης των μειονεκτικών περιφερειών και περιοχών, στον πρώτο πυλώνα. Πολλά, πολλές συζητήσεις έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες για τις προτάσεις για την πρόσθετη υποστήριξη για τους νέους γεωργούς. Το μέσο, το εργαλείο tool για τις μειονεκτικές ε, περιοχές και περιφέρειες ακόμα δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για αυτό το θέμα και θα έλεγα σε αυτό ακριβώς το θέμα θα πρέπει να συζητήσουμε και να σκεφτούμε τι πρέπει να γίνει ποιες θέσεις θα υιοθετήσουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί. Τις ορεινές περιοχές και τις μειονεκτικές περιοχές, αν θέλουμε να τις διατηρήσουμε για τη γεωργία, για τις γεωργικές δραστηριότητες, θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό πιο σύνετα και πιο αποτελεσματικά. Και για το θέμα της διαχείρισης κινδύνου συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το μέσο μόνο στο δεύτερο πυλώνα μπορεί να μεταφερθεί Εκεί έχει μεταφερθεί ώστε να μην έχουμε στον πρώτο πυλώνα κονδύλια τα οποία θα δημιουργούν πίεση και η άμεση επιδότηση, ας το πω έτσι, να μην συρρυκνωθεί από τον πρώτο πυλώνα. Το βρίσκω, ας το έτσι, ε, σαν ε, κατάσταση παράλογη. Από πλευράς προσέγγισης είναι περισσότερο λογικό τον κίνδυνο να τον καλύψουμε με την διασφάλιση εισοδήματος δράση στον πρώτο πυλώνα θα πρέπει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περάσει στον δεύτερο πυλώνα είναι συνετή ή όχι. Ή μήπως όχι μια παρόμοια λύση, αλλά να βρούμε τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την κατάσταση στα κράτη-μέλη όπου έχουμε παράπονα σε σχέση με την ε, κατάσταση για τον ε, η κατάσταση του πρώτου πυλώνα. Είναι ελεύθερη η επιλογή στα κράτη-μέλη αν θα το κάνουν αυτό βέβαια ή όχι, αλλά θα πρέπει να πετύχουμε μια πιο συνετή λύση σε σχέση με τα όσα προτείνει η Επιτροπή να μεταφερθούν στο δεύτερο πυλώνα. Και θα ήθελα να ζητήσω να ξαναπροβληματιστούμε για αυτά τα πράγματα, να βρούμε μια συνετή λογική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζωζέ μετά ο Λουίς Καπολασάν. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ευχαριστωμένος που σήμερα είναι εδώ ο Ρενέ Σουσόν και αντιπροσωπεύει τις ε, περιφέρειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε και είναι αλήθεια ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Ακούγοντας ε, την παρουσίαση, λοιπόν, λέω σκέφτομαι πως είναι κρίμα να είμαστε ακόμα στον τριμερή διάλογο ενώ θα μπορούσε να είναι τετραμερής και οι περιφέρειες θα μπορούσαν πολύ να μας βοηθήσουν σε αυτή την υπόθεση ιδιαίτερα στις χώρες όπου είναι πιο φοβισμένες και φοβισμένα τα κράτη και πιο μακριά από τις ανησυχίες του γεωργικού κόσμου. Απάντως προς αυτήν την ε, προοπτική θα πρέπει να ονειρευόμαστε του τετραμερούς διαλόγου. Δεν, πρέπει να, δεν θέλω να προβώ σε διαπιστώσεις, είναι σωστά όσον αφορά όλα αυτά που είπατε. Συμμερίζομαι βεβαίως στις θέσεις των περιφερειών και είναι σημαντικό νομίζω και θα, θα έπρεπε οι περιφέρειες στο πλαίσιο των προοπτικών της συζήτησης που θα έχουμε με το Συμβούλιο να μπορούν να περνούν το μήνυμά τους σε κάθε κυβέρνηση γιατί συχνά οι κυβερνήσεις είναι πολύ μακριά από τις διαπιστώσεις που κάνουν οι περιφέρειες. Το γεγονός ότι οι περιφέρειες λοιπόν διαπιστώνουν ότι πρέπει να ρυθμιστεί η ζήτηση και η προσφορά είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώ όμω αισθανόμαστε το αντίθετο και για τα θέματα τη δικαιοσύνη και τη κατανομή που είναι σημαντικά. Ε, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτά που ισχύουν σήμερα. Έχω τρει ερωτήσει να θέσω. Ε, τον εκπρόσωπο των περιφερειών. Δεν μιλήσατε για το ρόλο των μικρών ε, γεωρικών εκμεταλλεύσεων και θα ήταν σημαντικό να πείτε δύο λόγια για εδώ. Ε, φαντάζομαι ότι στο πλαίσιο της ε, τοπικής ανάπτυξης είναι κάτι το σημαντικό και επίσης το θέμα του πώς μέσα στο πρασίνισμα ε, διαρθρώνεται η δυνατότητα αποκατάστασης της αυτονομίας σε φυτικές πρωτεΐνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάλαβα πολύ καλά και ίσως εδώ να είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται να ε, ξεκαθαριστεί. Ε, δηλαδή πώς συνδέεται το θέμα του 7% ανάμεσα στις εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ε, τον, τον οικολογικό φόρο και την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία θα είναι κάτι πολύ δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ο Λουίς και μετά ο Μισελ Νταρντέν. Νταντάν, συγγνώμη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Σουσόν ανάμεσά μας. Μια εξέχουσα προσωπικότητα που σεβόμαστε πολύ για την πείρα που έχει όχι μόνο ως μέλους της Επιτροπής Περιφερειών, αλλά και ως πρώην κυβερνήτη ε, διαμερίσματος στη Γαλλία, νομάρχη. Και για αυτούς τους λόγους φυσικά οι απόψεις που μας διαβιβάζει είναι πολύ αξιόλογες και που τις προσέχουμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να πω για κάποιες από αυτές, σε σχέση με κάποιες από αυτές θα πρέπει να να μπορέσουν να εξευρεθούν απαντήσεις στην έκθεσή μου ιδιαίτερα για το θέμα της σύγκλησης ε, συνοχής εσωτερικής ή εξωτερικής. Και εδώ υπάρχει μια συμβατότητα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και τις προτάσεις, όσον αφορά την ταχύτητα που προτείνεται να ακολουθηθεί, πολύ μεγάλη όσον αφορά τα κράτη-μέλη και πολύ μικρή μεταξύ των κρατών μελών και γι' αυτό θα ήθελα να εισαχθεί μια πραγματική συνοχή, ας το πω έτσι, μειώνοντας όσον αφορά τους ρυθμούς ταχύτητας ώστε σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό να βρεθούν ανάλογα με τους ρυθμούς αυτούς οι σωστές ισορροπίες. Για το πρασίνισμα, το greening, θα πρέπει να βρούμε ε, σωστές αποφάσεις, σωστές αποφάσεις που θα στοχεύουν σε μια σωστή ισορροπία και για την πρόταση να επαναπεριφερειοποιηθούν τα μέτρα για το πρασίνισμα αντιμετωπίζουν κάπως, ας το πω έτσι, εμπόδια που ε, δημιουργούν δυσκολίες για την εφαρμογή τους. Μια και είναι ατομικές οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις και εκείνοι που παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτές είναι ατομικά οι γεωργοί και αντίστοιχα, αντίθετα, έχουμε σε σχέση με κάποιες πρακτικές για το περιβάλλον ένα άλλο διαφορετικό ευρύτερο πλαίσιο, δεν ξέρω πώς μπορεί ένας γεωργός να την χάνει της υποστήριξης ε, για την ε, εκμετάλλευσή του και να εξετάζονται σε άλλη κλίμακα για άλλους ε, ιδιοκτήτες τα περιβαλλοντικά μέτρα. Θα πρέπει και εδώ πάλι οι βέλτιστες προϋποθέσεις να ισχύουν ώστε να μην υπάρχει τέτοιος κατακαιρματισμός. Θα πρέπει αυτό να αντανακλάται επαρκώς. Αυτό είναι ένα εμπόδιο που δύσκολο καθιστά να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Θα έχουμε όμως σίγουρα ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα τους επόμενους μήνες μέλλον. Άλλη δυσκολία, άλλο θέμα με το οποίο όμως συμφωνώ είναι ένα άλλο θέμα όπου ο δικός μου προβληματισμός αντιμετωπίζει και εκεί κάποιες, κάποια προβλήματα είναι το θέμα των νέων εισαγωμένων. Εδώ για τους νέους εισαγόμενους στη Γεωργία, όχι μόνο νέους αλλά και άλλους, τίθεται πρόβλημα Δηλαδή να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι κινήτρων, να μπορούν να, βρούνε, να, να βρούμε έναν ορισμό για το τι είναι ένας νέος γεωργός. Γιατί ανοίγεται έτσι πόρτα και παράθυρο αν δεν υπάρξουν σαφείς ορισμοί για απάτες και καταχρήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τύχει σε βάθος προβληματισμού για να, να, να μην καταλήξουμε μια καλή ιδέα, μια καλή αρχή να υπονομεύεται, να μην λειτουργεί στην πρακτική. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις που ε, σε σχέση με την δική μου έκθεση είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια συνεδρίαση με την Επιτροπή των Περιφερειών. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας ώστε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που τώρα ξεκινά για αυτά τα θέματα αυτών των εκθέσεων να συζητήσουμε περισσότερο σε βάθος και να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε προτάσεις στο μέτρο του εφικτού. Ευχαριστώ. Grazie Luis. Michel E poi... Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή από την Επιτροπή των Περιφερειών για αυτά που μας είπε. Αναρωτιέται αν ακούγεται. Ακουγότανε, αλλά αλλάζει μικρόφωνο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω, επαναλαμβάνει ο μιλητή, τον εισηγητή για τόσα μας είπε. Από την άλλη βέβαια λυπάμαι που η παρέμβαση αυτή γίνεται αφού εμείς έχουμε ετοιμάσει την δικιά μας έκθεση. Βέβαια η Επιτροπή των Περιφερειών, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Κάπουλος Σάντος, απαντήσεις υπάρχουν στις προτάσεις τροποποίησης που έχουμε υποβάλει. Για να αλλάξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε κάποιες παρατηρήσεις μας να ληφθούν υπόψη. Για αυτά που ακούσαμε τώρα, έχω τρει-τέσσερι παρατηρήσει ή ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα για την κοινή οργάνωση αγορών. Σημείωσα την παρατήρηση τη Επιτροπή των Περιφερειών που ε, λυπάται για την εξαφάνιση διαφόρων ε, μέτρων που υπήρχαν μέχρι τώρα. Όμως δεν κάνει πρόταση για νέα μέτρα, ώστε να υπάρξει αυτή η ρύθμιση των αγορών. Υπάρχουν? Αν υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Από την άλλη, θέλω να ακούσω κάποιες διευκρινήσεις για αυτά που λέτε όσον αφορά τον ρόλο των περιφερειών στο δεύτερο πυλώνα. Η Επιτροπή των Περιφερειών πώς το βλέπει αυτό το θέμα. Και έρχομαι και στη διαχείριση του κινδύνου. Συμφωνώ με την ανάλυση που κάνετε. Δεν έχει κλείσει η συζήτηση εξάλλου με τον εισηγητή, ακόμα και αν έχει μείνει στο δεύτερο πυλώνα το θέμα, πάντα μπορεί να υπάρξει κάτι και στον πρώτο. Τέλος, για τους νέους γεωργούς. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δηλαδή πρέπει να χαίρει βοήθειας από το κράτος οποιοδήποτε ε, ξεκινήσει μια τέτοια δραστηριότητα, ό,τι ηλικία και αν είναι. Θέλω όμως να βάλω μια μικρή απόχρωση. Όταν κάποιος στα 25, στα 30 καθίστεται στην ε, Ήπεθρο, δεν έχει τα χρήματα για να αγοράσει μια παλιά ισχυρή εγκατάσταση και γι' αυτό χρειάζεται την ενίσχυση. Αυτή χρειάζεται δηλαδή μεγάλα κεφάλαια. Ενώ όταν στα 40, 45 ή 50 εγκαθίσταται κάποιος και να ξεκινάει μια τέτοια δραστηριότητα, θα έχει κάποιο κεφάλαιο στην πάντα ή τέλο πάντων μπορεί να το έχει για να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Όχι πάντα. Δεν μπορούμε φυσικά να μιλήσουμε για ατομικά διάφορες περιπτώσεις, μιλάω γενικά. Αν θέλετε το συζητάμε και παρετέρω. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μισελ. Τέλος. Άγνιου. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν θυμάμαι να αναφέρετε την επιμονή στο ότι οι γεωργοί θα πρέπει να καλλιεργούν τρία είδη. Στη Βρετανία το θεωρούμε αυτό πολύ άβολο, καθόλου απαραίτητο. Δεν θα πετύχει τίποτα απολύτω για το περιβάλλον. Περισσότερα ε, κόσμος θα βρεθεί στο δρόμο και στις ε, ρώσιμες γέζε λόγω του αυξημένου αριθμού ανθρώπων που θα πρέπει να ελέγχουν. Ε, έχω βρει κάποιους τρόπους. Το ένα είναι να μειωθεί ε, σε δύο είδη καλλιέργεια. Το τρίτο είναι να θεωρείται η συμμετοχή σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα ως μια καλλιέργεια και έπειτα να αυξηθεί το γελία χαμηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σχετική βοήθεια. Τα σχόλιά σας παρακαλώ θα ήθελα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Άγνιου. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή Ρενέ Σούσο και ευχαριστώ τον και εγώ που είναι σήμερα εδώ για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα βασικά ερωτήματα που ετέθησαν. Αν δεν σας δώσω όλες τις απαντήσεις ε, σήμερα, Πάντως θα είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω με τους εισηγητές ε, που το θέλουν. Ε, τώρα, για την ε, χρηματοδότηση είπα σαφώς, ακόμα και αν ε, δεν επέμενε και πολύ, αυτό που προτείνει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή 425,6 δις ευρώ, είναι το μίνιμουμ, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, αν μιλήσω ως Γάλλος, Είμαι από αυτούς που λυπούνται που η προηγούμενη γαλλική κυβέρνηση ζήτησε να μειωθεί η συμβολή της Γαλλίας, ε, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές δυσκολίες να διατηρήσουμε πολιτικές πολύ βασικές για την ΚΑΠ και για την, και την πολιτική συνοχή. Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι σαφής ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα τις μειονεκτούσες περιοχές, ε, τις ορεινές περιοχές, ε, εμείς ε, θελήσαμε πολύ να τους λάβουμε υπόψη ε, και θα έπρεπε να απομακρυνθούμε από μια τεχνοκρατική προσέγγιση, να πάψουμε να θεωρούμε ότι οι δύσκολες ζώνες, οι ορεινές περιοχές είναι ένα βάρος, ένα φορτίο. Στην πράξη, στην πραγματικότητα, στη σημερινή κοινωνία αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία. Για δείτε όλα τα βουνά της Ευρώπης. Τι είναι δάση, πώς θα μπορούσε η Ευρώπη να ακολουθήσει πολιτική βιοπικιλότητα αν δεν ασχοληθεί με τα δάση. Οι πηγές μας, οι πηγές ε, νερού ε, ψηλής ποιότητας που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη στις ορεινές περιοχές. Έχουμε και μια επιτροπή για τη κεντρική οροσυρά της Γαλλίας και μάλιστα μόλις τώρα είδαμε ε, μαζί με αυτή την επιτροπή ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ορεινές περιοχές και εκτός από τη Γεωργία που είναι βρίσκεται στην καρδιά. Για το σύνολο δεν μιλάμε της ε, κοινωνίας και διαπιστώνουμε έτσι ότι η εμπορική αξία αυτών των διευκολύνσεων είναι πολύ μεγάλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπολογιστή. Τώρα αρχίζει να γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή πια να θεωρούμε τις μειονεκτούσες περιοχές ως βάρος, ως ε, κάτι το οποίο είναι δαπανηρό, αντίθετα πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι το οποίο μας δίνει πολύ σημαντικούς πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και βεβαίω θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον κύριο Ντόρφμαν για αυτό το θέμα. Για την εγκατάσταση. Ναι, βεβαίως θα πρέπει να γίνει αυτό, αλλά αν έχουμε εισάγει εδώ τον, τους νέο εγκατασταθέντες, έχουμε περιλάβει εδώ τους άνω των 40 ετών. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια και θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τον ενεργό Γεωργό. Δεν το συζητήσαμε, αλλά ε, από τη στιγμή που υπάρχει ένα ποσοστό εισοδημάτων εκτός της ε, γεωργίας που είναι σημαντικό πέρα από 10.000 ευρώ μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι δραστήριος αυτός ο ενεργός αυτός ο γεωργός. Όχι, κατά τη γνώμη μας. Ε, κάποια κράτη θεωρούν ότι ο ενεργός γεωργός θα πρέπει να φεθεί στο δικό του ορισμό. Εγώ νομίζω πως είναι κάπως επικίνδυνο αυτό γιατί πρέπει όλα ένα και περισσότερο να διαχειριστούμε την διαφορετοποίηση της γεωργίας, ναι, α, α, αυτό εντάξει, αλλά το να αφήσουμε να ορίσουν από μόνοι τους ε, τους ενεργούς ε, γεωργούς, όχι. Για τα όσα είπε ο Ζωζίποβέ, τον... και εκεί θελήσαμε να τα συμπεριλάβουμε αυτά, αν και κάποιες φορές ήθελαν να εξαφανιστούν αυτέ οι καταποκοπήν ενισχύσει στι μικρού στις μικρές εκμεταλλεύσεις, εμείς θεωρήσαμε ότι μια βοήθεια χιλίων ευρώ μάλλον κάτω από τα χιλιά ευρώ δεν χρειάζεται να ελέγχεται. Άμα δούμε τον όγκο των ενισχύσεων που παίρνουν οι εκμεταλλεύσει, ιδιαίτερα στι νέε είναι θα δούμε ότι οι περισσότεροι είναι κάτω από το όριο των χίλιων ευρώ. Για τον τρόπο ελαστικής εφαρμογής αυτών των μέτρων, το 30% και το 7% των οικολογικών επιφανειών. Καταρχήν, τις πρωτεΐνες τις ζητάμε. Το πρόγραμμα για τις πρωτεΐνες τις ζητάμε και το περιλαμβάνουμε στο 30%. Δεν το είπα, αλλά είναι μέσα στην πρότασή μα, στη γνωμοδότησή μα ξεκάθαρα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα για τις πρωτεΐνες και κάθε φορά που θα γίνεται λόγος για τις καλλιέργειες των πρωτεϊνών θα πρέπει φυσικά να λαμβάνονται υπόψη. Ε, καθώς επίση θεωρούμε ότι τα μόνιμα βοσκοτόπια θα πρέπει α, α, αυτόματα να λαμβάνονται υπόψη. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη φάση, πώς διαχειριζόμαστε το 30% και το 7% πάντα συνεχίζοντας τις ατομικές πληρωμές. Όλα εξαρτώνται από το τι θα επιλέξει το κράτος ως τρόπο διαχείρισης. θα είναι ένας εθνικός τρόπος διαχείρισης ή άρθρο 20 περιφερειακής διαχείρισης. Αν είναι σε εθνικό επίπεδο το, το, το σύστημα που προτείνουμε, Δηλαδή, οι συμβάσει εταιρική σχέση ανάμεσα σε μια ομάδα γεωργών αναλεκάν παραγωγή και την ε, αρχή διαχείριση. Είναι δύσκολο είναι το κράτο γιατί πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι. Ενώ είναι πολύ εύκολο να επιλέξουμε την περιφερειοποίηση, γιατί οι περιφέρειες στο δεύτερο πυλώνα είναι παντού σε συγχρηματοδότηση. Παντού σε συγχρηματοδότηση. Στον πρώτο πυλώνα για την ώρα δεν παρεμβαίνουν. Η Κομισιόν ανοίγει τη δυνατότητα να μπορούν να παρέμβουν. Για μας αυτή είναι η λύση. Η λύση γιατί έχουμε έτσι διαχείριση του πρώτου και του πρώτου πυλώνα σε τοπικό επίπεδο, ε, εδαφικότητα και αυτά τα μέτρα πρασινίσματος. Η Ένωση φτιάχνει ένα κατάλογο πιθανών και, ε, καλλιεργιών και παραγωγών και στη συνέχεια αφήνουμε κάθε περιφέρεια μέσα σε συμβάσεις που κάνει με τους γεωργούς για μια συγκεκριμένη λεκάνη παραγωγής να επιλέξει. Ο έλεγχος της ε, περιφέρειας γίνονται, γίνεται έτσι από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρώπη. Δεν είναι πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι πλήρως ή μερικώ είμαστε αρχή διαχειριστική για τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία και για το ΦΕΝΤΕΡ διαρκώς και συστηματικά είμαστε στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης. Δηλαδή λίγο παραπέρα αρκεί να πάμε για την εφαρμογή του, του, των συμβάσεων ώστε να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε αυτά πολύ ελαστικά. Αν θέλουμε τα ίδια μέτρα να εφαρμοστούν παντού στο επίπεδο της Ευρώπης, ε, θα ξέρουμε τι θα γίνει. Πολλές μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις θα εξαφανιστούν γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν. Ε, το κλειδί της μελλοντική γεωργικής πολιτικής είναι το κατά πόσο θα έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στην ε, μεγάλη ποικιλία των εκμεταλλεύσεων. Χρειαζόμαστε όλες μας τις εκμεταλλεύσεις. Το λέει και η Κομισιόν. Α, πρέπει να έχουμε και τον τρόπο να πετύχουμε. Και για να μπορέσουμε να πετύχουμε πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ομοιόμορφα μέτρα διαχείρισης. Να πάμε πιο κοντά στην αγρονομική πραγματικότητα και την ανθρώπινη πραγματικότητα της κάθε εκμετάλλευση. και γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που όλο ένα και ε, μας λέει η Ευρώπη, στην πράξη δεν τα καταφέρνει τόσο καλά. Τρία επίπεδα λοιπόν ε, μπορώ να, το, να εξηγήσω και ακόμα περισσότερα σε άλλο πλαίσιο. Παρέλειψα μια σημαντική ερώτηση για τα εργαλεία ρύθμισης του του κυρίου Νταντά. Είπαμε ότι χρειάζεται ρύθμιση, αλλά ότι δεν έχουμε αρκετή, αρκετή ακτίμηση του αντίκτυπου της κατάργησης των ισχυών των μηχανισμών. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, αλλά όχι αρκετά εις βάθος. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της κατάργησης της ε, γαλακτοκομικής ποσότητας, για παράδειγμα, για τις εκμεταλλεύσεις των μειονεκτούσεων περιοχών. Δεν έχω ε, τα στοιχεία, αλλά έχω μάτια και βλέπω και από αυτιά και ακούω. Και βλέπω ότι η εξαφάνιση των γαλακτοκομικών παραγωγών στις ορεινές περιοχές εξαφανίζεται ταχύτατα, αν δεν γίνεται μετατροπή τους σε τυριά με με προέλευση, με συγκεκριμένη ονομασία προέλευση. Ξαφανίζεται πολλέ φορέ ολόκληρη η γαλακτοκιμική παραγωγή, γιατί ο κτηνοτρόφο που κάνει 150 λίτρα, 150.000 ε, λίτρα στο, στο βουνό, ε, είναι σε ανταγωνισμό με ε, γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις τεράστιες που φτιάχνουν ε, τόνους. Πριν να προτείνουμε λοιπόν άλλα εργαλεία ρύθμισης, πρέπει η Ευρώπη να κάνει συγκεκριμένες μελέτες, όχι μόνο απλά μακροοικονομικές, αλλά περιφέρεια, ε, για να δει ποια είναι, <coughs> ποιες είναι οι επιπτώσεις. Εγώ λέω ότι πρέπει να καταργηθούν, ναι, αλλά λέω επίσης ότι όταν είπα τις τις εισάγουν και η Ευρώπη τις καταργεί, Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει, το οποίο δεν έχουμε σωστά μετρήσει. Το 84 όταν εγκαταστάθηκαν, όταν εισήχθησαν οι ποσοστώσεις δεν έγινε καλά κατανοητό, πάντως σίγουρα ε, ήταν, επέτρεψε να προσαρμοστεί η παραγωγή και κατανάλωση και επέτρεψε και έσωσε τη γαλακτοκομική παραγωγή αυτό το σύστημα από πλήρη εξαφάνιση στις δύσκολες περιοχές. Και τότε εγώ ήμουν υπουργό. Γι' αυτά λέω δεν πρέπει να προσέξουμε, να προσέξουμε πριν να αλλάξουμε τις ισχύουσες διατάξεις και πάλι δεν μπορώ παρά να πω ότι μετά στη συνέχεια θα μπορέσουμε να λάβουμε τα πιο κατάλληλα μέτρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά μιλάμε για πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Είναι αλήθεια ότι οι τοπικέ αρχέ έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Υπογραμμίσαμε και όλο ιδιαίτερω οι περιφέρειε ότι δεν μπορούμε απλά να είμαστε οι συγχρηματοδότε, οι τραπεζίτε του δεύτερου πυλώνα τη ΚΑΠ, αυτό που είμαστε δηλαδή τη στιγμή έρχονται και να γράφουμε μόνο τα, επιταγέ. Πρέπει να έχουμε το συνολικό, τη συνολική εικόνα, να υπάρχει συνοχή, γιατί η Ευρώπη λέει ναι, κοινό στρατηγικό πρόγραμμα, να υπάρχουν ε, οι συμβάσει εταιρική σχέση, να, να είμαστε συνδεδεμένοι με όλα αυτά για να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και να ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα διαφοροποιημένη γεωργική πολιτική χωρί να πέφτουμε σε ε, βαριά συστήματα. Άλλη λύση εγώ δεν βλέπω από την περιφερειοποίηση της ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σούσον. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Όντω τώρα έμειναν δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη, συνάδελφοι το 8 και το 9, που είναι δύο εκθέσεις που ε, φροντίζει η Σάντρα Καλνιέτα που όμως ψηφίζει σε άλλη επιτροπή. Πέντε λεπτά διάλειμμα λοιπόν όταν θα έρθει πίσω η Καλνιέτα.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 η Σάντρα Καλνιέτε επανήλθε, οπότε μπορούμε να δούμε τα σημεία 8 και 9 που είναι τα τελευταία δύο που μας έχουν μείνει στην ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου ωστόσο σύντομα να χαιρετήσω θερμά και να καλωσορίσω την ομάδα ε, του προσωπικού του Αμερικανικού Κογκρέσου από την Επιτροπή Γεωργίας. Να ευχαριστήσω επίσης το Ίδρυμα Πέτερσμαν καθώς όπως ξέρετε συνάδελφοι ε, μια ανταλλαγή ανάμεσα στο προσωπικό της δικής μας Επιτροπής Γεωργίας και των ε, ομολόγων τους στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία γιατί έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε τον ε, ε, διατλαντικό διάλογο κυρίως σε αυτή την περίοδο που όπως γνωρίζετε συζητά το Αμερικανικό Κογκρέσο τη μεταρρύθμιση του Pharma Bill του νόμου περιγεωργίας, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δική μας μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Να σας καλωσορίσω λοιπόν κάποιοι από τους βοηθούς μας μαζί με αυτή την ομάδα των Αμερικανικών συναδέλφων είναι για τους ευχαριστώ για τη δουλειά τους και προχωράμε με το σημείο 8 η θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία. Συντάκτρια γνωμοδότησης ε, είναι η Σάντρα Καλνία. Ε, 24 Απριλίου θα τα ε, αποφασίσαμε ότι θα δούμε από κοινού αυτά τα προγράμματα το ορίζον 2020 δηλαδή. πρώτη γνωμοδότηση αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο στο σύνολό του. Το δεύτερο τμήμα αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά την Επιτροπή Γεωργίας. Το βασικό ζήτημα για την Επιτροπή Γεωργίας είναι το ίδιο. Δηλαδή ποια είναι οι προτεραιότητές μας. Αγαπητή Σάντρα, έχεις το λόγο. Ε, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ε, ε, ήθελα να πω ότι σε σχέση με Έπρεπε πιο πριν ε, να απασχοληθώ στην ε, ήμουνα με ανηλυμένε υποχρεώσεις σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και σας δω συγγνώμη. Ξεκινώ ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες τους, προετοιμάζοντας ε, το έγγραφο για τον ορίζοντα 2020. Επειδή αυτή η πρόταση φυσικά στοχεύει σε αυτές τις βελτιώσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα και τη βελτίωσή της. Είναι η πρώτη φορά όταν έχουμε θέματα χρηματοδότησης που στοχεύουν για την έρευνα και την καινοτομία. Έχουμε κάποιους τομείς που ομαδοποιούνται. Ο ορίζοντας 2020 στοχεύει άμεσα στην προαγωγή, στην προώθηση επιστημονικών καινοτόμων πρωτοβουλειών και τη μετάφρασή τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες μια και αυτή η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις βελτιώνοντας και τη ζωή των πολιτών μας ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Στόχος είναι να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος, η γραφειοκρατική επιβάρυνση, απλουστεύοντας τους κανόνες του παιχνιδιού και τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας ότι υψηλά προσοντούχα άτομα, επιστήμονες θα συμμετέχουν στην καινοτομία και στην έρευνα και θα συμμετέχουν επίσης εκείνες οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να υλοποιήσουν αυτές τις καινοτόμες δράσεις. Όπως τόνισα, στην, υπογράμμισα στην γνωμοδότησή μου, επικεντρώθηκα σε εκείνα τα θέματα τα οποία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και συνδέονται τις περισσότερες φορές με τη Γεωργία. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας έλαβα υπόψη και σημείωσα τις ανησυχίες και τα μελήματα των συναδέλφων Υπάρχει η δυνατότητα η επιστήμη, η επιστήμη να προτείνει πολύ σημαντικές ιδέες που πολλές φορές δεν υλοποιούνται στην πραγματική ζωή διότι δεν εμπλέκεται η ίδια η κοινωνία, δεν φτάνουν τα μηνύματα στους αποδέκτες, στους πολίτες. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να επανορθώσουμε αυτή την έλλειψη πληροφόρησης να διαχέονται οι πληροφορίες και να υπάρχει ένας σε διάλογος μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των άλλων εμπλεκόμενων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και υλοποίησης των προγραμμάτων ώστε να εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράδειγμα κάνοντας λόγο για τους δικούς μας τομείς ενδιαφέροντος για τη γεωργία, διάφορες ενώσεις και συλλόγους γεωργών έχουν τεράστια πείρα και πολύ μεγάλη πρακτική γνώση και θα ήταν ανεκτήμητο να μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτόν τον διάλογο οι γεωργοί και οι εμπλεκόμενοι από αυτόν τον διάλογο με τους επιστήμονες και την καινοτομία. Ορίζοντας 2020 στοχεύει στο να πετύχουμε η κοινωνία να, εφοδιάζει, να εφοδιάζεται με υγιεινές τροφές και ασφαλείς τροφές και τρόφιμα. Μέσα στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή εκφράσαμε επανειλημμένα τις ανησυχίες μας για την αύξηση της ζήτησης τροφίμων και η αύξηση αυτή θα επιταθεί, θα ε, αυξηθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες. Είναι επιτέλους τώρα η χρονική στιγμή να προβληματιστούμε και να δούμε πώς θα καλύπτουμε τις διατροφικές μας ανάγκες, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να ξεπεράσουμε. Πιστεύω ότι πολλοί οργίζονται και δίκαια εξοργίζονται επειδή μεγάλο ποσοστό των παραγόμενων τροφίμων πάνε στα σκουπίδια και δεν, ε, δεν μπορεί να υποφεληθεί ο κόσμος ε, από την, ε, στη διατροφή του από αυτά. Πρέπει να βρούμε πρακτική επίλυση αυτού του προβλήματος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε τα τρόφιμα τα οποία καταλήγουν στους νεκέδε. Υπάρχει και ένα σχέδιο λοιπόν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση και του γραφειοκρατικού βάρους να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 7 Ιουνίου. Και πραγματικά ελπίζω, ευελπιστώ ότι οι συνάδελφοι θα δραχθούν της ευκαιρίας και θα είναι σε θέση να υποβάλουν τέτοιου είδους θετικές προτάσεις ή και τροπολογίες. Λόγω των προβλημάτων όσον αφορά χρονοδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα και τη συναντήσεις μας δεν είχα ευκαιρία να συνέρθω και να διαβουλευτώ με τους κοιόδης εισηγητές. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι θα επανέλθω και θα κερδίσουμε το χρονικό διάστημα που χάσαμε σε σχέση με τις ε, τροπολογίες. Πρέπει να τις εξετάσουμε με καλό θετικό τρόπο για να υπάρξει ισορροπημένη άποψη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ε, και τώρα έχει το λόγο ο Ζωζέ Μποβέ. Ναι, κυρία Ισηγήτρια, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και είναι αλήθεια ότι τα όσα λέτε έχουν, ε, είναι λογικά. Και όταν διαβάζουμε την πρόταση της ε, Κομισιόν ε, πραγματικά ανησυχούμε γιατί είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα ε, από τις γεωργίες. Σαν να θέλουν να κάνουν ένα νέο δώρο σε ένα λόμπι το οποίο έχει κάνει πάρα πολλές ζημιές, έχει ταπανίσει, σπαταλήσει χρήματα σε προγράμματα που έχουν φυτρώσει από εδώ και από εκεί και την ιδέα της βιοοικονομίας και αυτή δεν την καταλαβαίνω. Η Γενική Διεύθυνση Έρευνα ε, χρηματοδοτεί προ προβλήματα τα οποία δεν είναι η πρώτη ανησυχία τη Γεωργία αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι από το 82 500 ε, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν ε, για αυτά τα θέματα και 200 εκατομμύρια ευρώ στις 10, τα 10 τελευταία χρόνια. Διόλευ καταφρόνουν τα ποσά με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν ώστε να γλυκάνουν το χάπι το, στο, για τον Ευρωπαίο πολίτη λέγοντας ότι ήταν ε, καλοί οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Ήταν το End Trans Food ε, το πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει τώρα πρέπει να πούμε στην ουσία, αυτά είπε και ο κύριος Σιόλος ε, και η κυρία Κόν και Ντεγκάρντ, ότι δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις νέες ε, προβληματικές που είναι ε, το θέμα της βιοπικιλότητας, το θέμα της σημείωσης του κόστους για τους γεωργούς, το κόστος παραγωγής με άλλες ε, ε, γεωργικές πρακτικές, ώστε να είναι πιο οικονομικές και πιο αυτόνομες. Και αυτό λέει άλλωστε και το πρόγραμμα SCAR που γνωρίζετε, της Μόνιμης Επιτροπής για τη Γεωργία και την Έρευνα, που αυτή τη στιγμή ε, δείχνει και λέει, τονίζει ποιες είναι οι αλλαγές που χρειάζονται. Λέει επίσης ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν οι ιστορικές γνώσεις, η τεχνογνωσία των, Γιωργών γεωργών βασικά σε όλα αυτά. Όλα αυτά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι στην καρδιά του... της πολιτικής μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς μόνο μία γνωμοδότηση κάνουμε, αλλά ο γεωργικός προπολογισμό στο πλαίσιο της, ε, του ερευνητικού προπολογισμού θα πρέπει να μεταφερθεί στη γεωργία και να εσωματωθεί στον τομέα της γεωργίας έτσι ώστε να είναι πολύ πιο μάλλον κάτι τέτοιο είναι κατά γνώμη πολύ πιο σκόπιμο από το να τα αφήσουμε στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Μας περιπτώσει αυτή είναι η γνώμη μου και σας ευχαριστώ. Για την πρόεδρος Πόλσον. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά επίσης ε, και την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που επετέλεσε και παρουσίασε. Συμφωνώ απόλυτα όταν αναφέρεται ότι είναι θετική η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για βελτιώσεις. Είναι σαφές ότι ο ορίζοντας 2020 είναι ένα τεράστια σημασία μέσο, ένα εργαλείο για την καινοτομία και την έρευνα όσον αφορά την γεωργία, την δασοπονία, ή και γενικά όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες της Γεωργίας. Για την Επιτροπή Γεωργίας στην Ευρωβουλή είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον τρίτο πυλώνα, να επισημάνουμε αυτή τη σπουδαιότητα του τρίτου πυλώνα, δηλαδή τον εφοδιασμό με τρόφιμα για θέματα διατροφής, ε, την κτηνοτροφία και άλλα συναφή θέματα έχει τεράστια σημασία να προσπαθήσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου να προβληματιστούμε και να δούμε σε ποια σημεία η πολιτική μας για τη γεωργία και η έρευνα πραγματικά συνδέονται, μπορούν να συνδεθούν και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ώστε οι γνώσεις των γεωργών στην γεωργία, στους τομείς τους γεωργικούς θα μπορέσουν να δώσουν θετικά αποτελέσματα και να τα μεταλλευτούμε όλα αυτά τα στοιχεία στο βέλτιστο, με το βέλτιστο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό στις γνώσεις αυτές να είμαστε με θετικό πρόσημο να προχωρήσουμε ώστε η έρευνα να μην αναφέρεται μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να μην μπορεί να επεκταθεί πέρα από αυτό ή πέρα από αυτήν. Έρευνα ακόμα και σε σχέση με την κτηνοτροφία και την, τα θέματα ε, εφοδιασμού με τέτοια προϊόντα. Δεν είναι απλό το εγχείρημα. Δεν πρέπει μόνο για μια μικρή συγκεκριμένη ομάδα να ισχύουν όλα αυτά, αλλά για όλους που έχουν και εμπλέκονται σε αυτή την πρακτική, ε, ας το πω έτσι, συνιστόσα για θετικά αποτελέσματα. Αυτά πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής μας λοιπόν και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Καινοτομία και τις Τεχνολογίες. Αυτό είναι κάτι που και στο πρόγραμμα για τον ορίζοντα 2020 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχει εδώ κάτι όπου αναφέρεται, όπου λέγεται ότι οι γνώσεις γνώσεις ανά ομάδες, ανακατηγορίες καινοτομίας. Γίνεται η προσπάθεια να ομαδοποιηθούν, να συνδεθούν διαφορετικοί γνωστικοί τομείς μεταξύ διαφορετικών φορέων, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων τέτοιων φορέων, ώστε οι βέλτιστες ικανότητες και επιδόσεις να επιτυγχάνονται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ομάδα που στόχος της είναι τα τρόφιμα, η αλυσίδα τροφίμων, η τροφική αλυσίδα να εξετάζεται σε βάθος. Αυτό είναι το θέμα αυτής της ε, εξειδικευμένης ομάδας. Και εμείς από πλευράς της ομάδας μας θα υποβάλουμε, θα καταθέσουμε συγκεκριμένες τροπολογίες που θα κάνουν λόγο για αυτά τα θέματα. Άμεση διασύνδεση μεταξύ των θεμάτων των δραστηριοτήτων της γεωργίας και της δασοπονίας για το επόμενο πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πτυχή που πιστεύω ότι είναι σημαντική για την μελλοντική κατεύθυνση για τους προσανατολισμούς της πολιτικής έρευνας. Πρέπει κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποστηριχθούν Μέχρι σήμερα διατίθενται υπερβολικά πολλά κονδύλια σε μεγάλα θεσμικά όργανα ή μεγάλες, ε, ε, μεγάλους φορείς και έτσι ε, εγκλωβιζόμαστε σε ένα, σε ένα ελεφάντινο πύργο ε, σε, ένα στεγανά που δεν ε, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε απήχηση ευρύτερη. Πρέπει λοιπόν αυτό να δούμε, την πρακτική εφαρμογή. Έχουμε και το θέμα της ε, διασπάθησης τροφίμων. Είχαμε και το θέμα της των δυνατοτήτων για την γεωργία όσον αφορά το νέο πρασίνισμα, μια νέα πράσινη επανάσταση. Και όλα αυτά συνδέονται φυσικά και με τη γενετικά τροποποιημένη τεχνολογία. Όλα αυτά όμως έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε αδιέξοδο. Πρέπει να αυξηθούν οι πόροι ε, όσον αφορά την έρευνα, να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί και να έχουμε καλύτερες επιδόσεις στην εκμετάλλευση των πόρων. Να δούμε περισσότερο και τη συνιστόσα της αηφορίας, την αηφόρο ανάπτυξη και να δούμε ποια είναι τα καλύτερα μέσα ώστε να προαχθεί μια γεωργία που με λιγότερο input όσον αφορά την εκμετάλλευση δηλαδή ορυκτών καυσίμων θα είμαστε πιο αποδοτικοί στις δράσεις μας. Αυτό πρέπει να πετύχουμε σε αυτή την αλλαγή προτύπου και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και κάποιες άλλες έννοιες ως ορόσημα προηγούμενα και σε άλλη συζήτηση αναφέρθηκε αυτό ότι στην Ευρώπη κάποιους τομείς για την έρευνα πρέπει να τους λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Έρευνα για τα φυτοκομικά προϊόντα, για τα φυτά. Έχει, έχει παραμεληθεί αυτός ο τομέας και πρέπει στοχοθετημένα να ενταχθεί ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι μακροπρόθεσμα θα εξαρτώμαστε πάντα από εισαγωγές σόγιας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Jim Nicholson. Ευχαριστώ Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εκθεσή της για τα δύο αυτά θέματα. Στην Επιτροπή αυτή έχουμε περάσει πολύ χρόνο να συζητάμε για τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ίσως όμως δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με τη βελτίωση της κατάστασης του πλαισίου της έρευνας. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε αυτή η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια για τον γεωργικό κλάδο και για όσους εξαρτώνται από αυτήν στην κοινωνία μας. Πρέπει να θερύνουμε τα πανεπιστήμια, τα γεωργικά Ινστιτούτα, με νέες ιδέες για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που μας έρχεται από ιδέες βασισμένες στην επιστημονική γνώση. Οι προκλήσεις που θα έχουμε και στο μέλλον θα είναι πολύ μεγάλες. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, για παράδειγμα, και όχι μόνο. Αυτή την ευκαιρία λοιπόν πρέπει να την δράξουμε και να την χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ο κόσμος πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται τις ποσότητες τροφίμων που σπαταλούνται στην Ευρώπη. Μπορεί να μιλάμε για το λοιμό στον κόσμο, αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μειωθεί η σπατάλη αυτή κατά 5% θα υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή. Τώρα για τις προτεραιότητές μας. Ένας από τους τομείς που πιστεύω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα για μας είναι η βιοπικιλότητα, η διαφοροποίηση. Γιατί όταν μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για 300-350 υπαλλήλους. Αλλά υπάρχουν και πιο μικρές. Με ένα άτομο, με δέκα άτομο. Στη Γεωργία Υπάρχει αυτό. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν, να βοηθήσουμε τέτοιου είδους επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλές ιδέες και τα κονδύλια να πάνε εκεί που υπάρχουν ιδέες. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ζωή των ανθρώπων της ε, υπαίθρου. Αυτό μπορεί να γίνει με νέες ιδέες. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε έρευνα για να έχουμε αυτές τις ιδέες. Εκεί όπου είναι και η καρδιά του κλάδου, στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τζιμ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τη Σάντρα Καλνιέτε. Είναι σημαντικό Α, για περιμένετε, γιατί ο Άγνιο ζήτησε το λόγο και μετά θα πω και εγώ δύο λόγια. Ναι. Άργησα λίγο, ναι, συγγνώμη. να δούμε πού μπορεί να υπάρχει συμφωνία. Εγώ συμφωνώ με τους πράσινους όσον αφορά την αρχή των ε, τροφίμων ε, των λιμάτων, αλλά πολλά από αυτά σπαταλώνται σε τρι... λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ας πούμε, τα ψάρια που απορρίπτονται, η υποχρέωση να πουετάν τα ψόφια ψάρια στη θάλασσα. Μα πόσο αυτό αποφελεί, γιατί το κάνουμε. Μετά έχουμε και τα απόβλητα, τα λίματα των σφαγίων θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν σε λιπάσματα για παράδειγμα, γιατί υπάρχουν πολλά ε, φωσφορούχα μέσα σε αυτά. Και μετά τα πόβλητα των, ε, από των εστιατορίων, τα λίματα, ναι, τα περισσέματα από τα εστιατόρια. Ε, αυτά τα βάζαμε, τα δίναμε στα γουρούνια. Τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το απαγορεύει αυτό. Γιατί όλα αυτά να τα πετάμε. Μάλιστα. Πριν να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, την κυρία Ρούτα, ε, θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Καλνιέτε γιατί λαμβάνει υπόψη το θέμα της ασφάλειας τροφίμων. Ε, δεν μπορούμε να μιλάμε υπόψη στα ερευνητικά μας προγράμματα για το μέλλον αυτά τα μεγάλα θέματα ε, για το αύριο. Δηλαδή πώς θα καταφέρουμε να αυξήσουμε το ευρωπαϊκό γεωργικό δυναμικό γιατί έχουμε σίγουρα ένα μέγα πρόβλημα έλλειψης τροφίμων στον κόσμο και η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει απ' έξω. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη συζήτηση και δίνω το λόγο στην Διευθύντρια της Επιτροπής, την κυρία Ρούτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας παρακολουθώντας τη συζήτηση. Είμαι η αρμόδια διευθύντρια για θέματα γεωργίας και έρευνας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε αυτή την έκθεση της κυρίας Κανιέτε και κυρίως ότι προσανατολίζεται στα κυριότερα θέματα όσον αφορά το πρόγραμμα για την έρευνα και αυτά που καλύπτει. Το ίδιο το ζήτημα του να προσπαθήσουμε καλύτερα να υποφεληθούμε από τα κονδύλια για την έρευνα και να στοχεύουμε σε καλές λύσεις για τα θέματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι μια καλή λύση και βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά του επόμενου προγράμματος πλαισίου που όπως ξέρετε αφορά και την έρευνα και την καινοτομία και όχι μόνο την έρευνα. Πράγματι λοιπόν επικεντρωνόμαστε με, ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη δράση στον τρόπο να υπάρξει η μεταφορά, η μετάθεση γνώσεων και πρακτικών ώστε να υποφεληθούν οι γεωργοί από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, της επιστημονικής έρευνας και με τους συναδέλφους μας στη Γενική Διεύθυνση για τη Γεωργία στην καινοτόμα εταιρική σχέση για την ε, έρευνα και τη γεωργία, αυτοί οι δεσμοί μπορούν να ενισχυθούν, να ενδυναμωθούν και οι παθητικές γνώσεις των γεωργών να λαμβάνονται υπόψη και να υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης με feedback μεταξύ γεωργών και επιστημόνων για να είμαστε πιο αποδοτικοί. Έτσι λοιπόν αυτή η έκθεση γνωμοδότηση εξετάζει ακριβώς, ε, στο, ε, βρίσκεται στο επίκεντρο των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν έχει μια ε, επιστημονική αξιόλογη αξία αλλά πρέπει να συνδεθεί και με την πρακτική εφαρμογή στις δράσεις για τη γεωργία. Σύμφωνο ότι πρέπει να μειώσουμε τη διασπάθηση τροφίμων, να μην πετάμε τα τρόφιμα στα σκουπίδια. Αυτό πρέπει να μειωθεί, πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η δράση. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που καταλήγουν στα, στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά πρέπει να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο για διάφορα απόβλητα, τα οποία δεν χρησιμοποιούμε, που θα μπορούσαμε όμως να τα εκμεταλλευτούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο. Ανέφερε ένας από τους προλαλήσαντες ε, τα απόβλητα των ε, ε, σφαγίων και τι θα μπορούσε να γίνει με αυτά. Αλλά παράδειγμα και για την έρευνα θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική των ασυνήθιστων λύσεων. Έχουμε ένα πρόγραμμα για την εκμετάλλευση ας το πω έτσι, του άνθρακα όσον αφορά τα απόβλητα. Παράδειγμα, την ανακύκλωση των πλαστικών. Τέτοιου είδου ασυνήθιστε ξεχωριστές λύσεις είναι κάτι το οποίο εξετάζουν οι επιστήμονές μας για να δράσουμε αποτελεσματικά. Και πέρα από αυτά για άλλες παρατηρήσεις που έγιναν από τους άλλους ε, προλαλήσαντες και τον αξιότιμο κύριο Αντιπρόεδρο για τη βιοοικονομία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η βιοοικονομία δεν είναι καθόλου ξένη και απομακρυσμένη από τη γεωργία. Αντίθετα βρίσκεται πολύ κοντά στις πρακτικές εφαρμογές ε, και στις ίδιες τις πρακτικές ε, της γεωργίας. Και ο όρος βίο προέρχεται από την βιολογία, όχι υποχρεωτικά από τη βιοτεχνολογία αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες δυνατότητες των βιολογικών πόρων με αηφορία, με αηφόρο τρόπο. Να χρησιμοποιούμε τους πόρους από τα εδάφη, την εκμετάλλευση των εδαφών, των δασών, στην δασοπονία. Να έχουμε την βέλτιστη χρήση τεχνολογιών ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, ώστε όλοι να μπορούμε να ε, εκμεταλλευτούμε στο βέλτιστο τους πόρους του πλανήτη χωρίς να τον λαιλατίσουμε. να εκμεταλλευτούμε λοιπόν ε, τους πόρους με αηφορία. Από την άλλη πλευρά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από άλλους, η εξάρτηση της Ευρώπης από τους ορυκτούς ε, φόρους, από τους ορυκτούς πόρους, τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να δούμε την εκμετάλλευση ευρωπαϊκών πόρων ως δυναμικού, βιομάζας και άλλων τέτοιων δυνατοτήτων. Να εκμεταλλευόμαστε αυτά για να έχουμε την παραγωγή που χρειάζεται, την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας μας. Και αυτό δίνει μια ευκαιρία για πολυμορφοποίηση των δραστηριοτήτων στις ε, αγρονομικές, αγροτικές δραστηριότητες. Θα έδιναν όλα αυτά θέσεις απασχόλησης ε, στον χώρο της υπαίθρου, προσφέροντας το εισόδημα για όσους θα εμπλεκόντουσαν. Ένα άλλο σημείο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ σημαντική υπόθεση αυτή. Βλέπουμε ότι ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλο και περισσότερο ε, την χάνουν υποστήριξη από ό,τι στο παρελθόν και πρέπει να υποστηρίζονται με κονδύλια, προγράμματα, σχέδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποκτούν μεγαλύτερη κλίμακα και μεγαλύτερη εμβέλεια και σε σχέση με τους, ε, ε, τη γεωργία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλο και περισσότερο ευδιάκριτο χαρακτήρα έχουν και συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Είναι σαφής λοιπόν η τάση και ο προσανατολισμός να βελτιωθούν οι δυνατότητες για την έρευνα όσον αφορά ε, την χρήση τους και από ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το οποίο τονίζετε εσείς ε, στην έκθεσή σας είναι σημαντικό. Η ανάγκη δηλαδή να υπάρχουν επαρκή κονδύλια θεμελιώδου ε, θεμελιώδους σημασία σε αυτό το σημείο. Αν δούμε το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης, συνειδητοποιεί κανείς ότι έχουμε λιγότερα από 2 δις ευρώ για ένα πολύ ευρύ πλαίσιο δράσεων που ξεκινά και καλύπτει από τα εδοφολογικά θέματα και την ανάλυση τους από την επιστήμη, γεωργικές πρακτικές και ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών ζητημάτων που καλύπτονται. Και μια και είναι τόσο διευρυμένο αυτό το πλαίσιο πρέπει και τα κονδύλια να επαρκούν σε ένα ευρύτερο, σε μεγαλύτερο βαθμό. Έχουμε σημειώσει όλες τις προτάσεις αυτές και σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για την κατανομή κονδυλίων για τη γεωργία και τη βιοοικονομία η πρόκληση που αντιμετωπίζεται έχει διπλασιαστεί πλέον, έχει πάρει διπλάσιες διαστάσεις. Η συζήτηση για τα κονδύλια στον προϋπολογισμό θα πρέπει λοιπόν αυτή την τάση να ακολουθήσει, να υπάρξει μια καλή παρακολούθηση όσον αφορά τα κονδύλια για τα, θέματα, τα επιστημονικά θέματα που συνδέονται με τη γεωργία ώστε να επαρκέσουμε, να υπαρκούμε από πλευράς κονδυλίων. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Οι συζητήσεις φυσικά θα συνεχιστούν και προσβλέπουμε στη γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρούτε και τώρα να ακούσουμε τα συμπεράσματα της Σάντρας Καλνιέτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλωσορίζω τις ε, παρατηρήσεις σας στο πλαίσιο του Horizon 2020. Ε, Είμαι έτοιμη για ανοιχτή και επικοδομητική συζήτηση, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε καλές συμβιβαστικέ ε, λύσεις αποδεκτές στην πλειοψηφία. Και έτσι να φτάσουμε σε μια καλή και ισορροπημένη γνωμοδότηση. Ωραία, σας ευχαριστώ όλους γιατί κλείσαμε έτσι τη συνεδρίασή μας για σήμερα το πρωί. Σας χαιρετίζω όλους και σας θυμίζω ότι η επόμενη θα είναι πάρα πολύ σημαντική στις 18 και 19 Ιουνίου. Οπότε οι εισηγητές μας θα παρουσιάσουν τις προτάσεις μας για την ΚΑΠ. Ευχαριστώ.